πολύ σημαντικό δυστυχώς το γεγονός και χρειάζεται να ρίξει μια ματιά και σε τέτοια πράγματα η Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε.